μας. Ε, αυτό να μην το ξεχνάμε. Η πρώτη ψηφοφορία τώρα. Μαλάουι και λοιπές αφρικανικές χώρες. Έχουμε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος. Δεν παραγραφώ 3 με την τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Το επόμενο αφορά τους τατάρους της Κρυμαίας και τους ηγέτες τους Τσιγκόζου Μέροφ και τον δημοσιογράφο Σέμενα. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το επόμενο αφορά την κατάσταση στις Μαλδίβες. Κοινή πρόταση ψηφίσματο από διάφορε πολιτικέ ομάδε. Το αρχικό κείμενο παραγραφού 5 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Τη παραγραφού 5 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Παραγραφός 8 τροπολογική παριθμών 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγωγός 14. Σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Είναι παραγραφό 15 δώσουμε το λόγο στον κύριο Τάνο, ο οποίο πρόκειται να μα εξηγήσει την προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Η πολιτική μα ομάδα θέλει να γίνει μια προφορική τροπολογία όσον αφορά την απάλληψη τη παραγράφου 15. Διότι από ό,τι μα υπηρεσίε εξωτερικέ ε, δράσει ότι είναι λανθασμένη αυτή η διάταξη και θέλουμε την διαγραφή τη. Την παράγραφο 15. Σας ευχαριστώ κύριε. Ποιο είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι αρκετή. Επομένως θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την αιτιολογική. Σι, κύριε Τάνοκο, έχετε πάλι το λόγο μας εξήγησε την προσφυγή τροπολογία. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, και εν προκειμένου ε, σύμφωνα με τόσο ε, μας είπε η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία ε, μας είπαν ότι πρέπει το, εκεί που λέει leader να βάλουμε former, πρώην ηγέτης γιατί δεν είναι πλέον ηγέτης. Πρόκειται για διόρθωση αυτού του πραγματικού περιστατικού. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι κατά της τροπολογίας της προφορικής τροπολογίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την ε, έκθεση της κυρίας Ματέρα για την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια. Και τώρα έχουμε την τελευταία μας ψηφοφορία αφορά την έκθεση Μπερζερών, σοφρονιστικά συστήματα και συνδικέ κράτηση. Το εναλλακτικό ψήφισμα του ΙΕΝΕΦ, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παραγωγός 7 το λογικό κειμένο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 12. Αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφορίας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Και τώρα ψηφίζουμε όλο το κείμενο μαζί με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα προχωρήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου.